Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ξεκινήσουμε αμέσως με τις ψηφοφορίες. Το πρώτο θέμα που θα ψηφίσουμε είναι η Παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών κατάργηση της οδηγίας 90-167 του Συμβουλίου. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Αγγιλέρα, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ίσως πριν να αρχίσουμε την ψηφοφορία να δώσω το λόγο στην κυρία Αγγιλέρα για να μας πει δύο λόγια. Ή προτιμάει αργότερα. Θέλει το λόγο τώρα ή προτιμάει αργότερα. Η κυρία Αγγιλέρα λέει ότι μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Έχουμε 401 τροπολογίες, 346 από τη δική μας Επιτροπή, οι υπόλοιπε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και υπάρχουν και αρκετές συμβαστικές τροπολογίες, 11 τον αριθμό. Ελπίζω να έχετε φέρει μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Τις συμβιβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ε, χάρη δεν θα ρωτάω κάθε φορά κατά και αποχές, μόνο υπέρ. Μην με παρεξηγείτε, απλώς για να επιταχύνουμε. Λοιπόν, περνάμε στη ψηφοφορία 41 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ διανατάσεως της χειρός, παρακαλώ, υπέρ τη τροπολογίας 41. Εγκρίνεται. Τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό τρόπο. Για την συμβαστική τροπολογία 7 άρχεται η τροπολογία. Κρατάει πιο πολύ η πρώτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας παρακαλώ. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 7. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 8. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 8. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 98. Στην τέταρτη σελίδα περνάμε κατευθείαν. Τροπολογία 98, Σάνι. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 98 παρακαλώ. Σάνι, διανατάσσεως χειρός. Εγκρίνεται η 98. Τροπολογία 99 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. 99. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 101 πρώτο τμήμα. Α, έχει αποσυρθεί το πρώτο τμήμα. Περάμε στην 102, η 101 έχει αποσυρθεί. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Α, 102, δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, διανατάσσεως της χειρός. 102, δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 103 του κυρίου Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 106. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Καταπίπτει. Τροπολογία 107. 107. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 107. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. 8. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Η τροπολογία 9 Τροπολογία 9. 9, γιατί 8 έχει καταπέσει, ψιθυρίζει ο γραμματέα. Εγκρίνεται η 9. 109 και 110. Ποιος είναι υπέρ της 109 μόνο, 109 μόνο. Ή 119 λέει τώρα ο πρόεδρος, Μπούδα και Ταντσίλα, εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα τέσσερα 130... Όχι, διορθώνει ο 136. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών 136 και 137. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται μάλλον. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Υπάρχει ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Κάποιος παρακαλώ να σταματήσει να ψηφίζει από το ΕΛΚ. Περισσεύει μία ψήφος του ΕΛΚ. Οπότε επαναλαμβάνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική 11. Τέλος, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 144, τον Αντρίου και Ντενανό. Ποιος είναι υπέρ της 144. Εγκρίνεται 144. 143. Ποιος είναι υπέρ. Okay, 100, επανάληψη της ψηφοφορίας για την 144. Ποιος είναι υπέρ με την 145 που είναι ταυτόσιμες. Το είχαμε ψηφίσει, εν πάση περιπτώσει ξαναψηφίζουμε. Εγκρίνονται. Τροπολογία 143. Ποιος είναι υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Πάμε στη 13. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 149. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 150 της κυρίας Κέστιγκερ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Περνάμε στην τροπολογία 160. Διανατάσεις της χειρός ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της 160. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 τώρα. Της συγγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 162 δεύτερο τμήμα. 162 δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της 162. 18. 163. 163 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 163. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής τροπολογίας 1. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 189. Σελίδα 8. Ποιος είναι υπέρ της 189, παρακαλώ σηκώστε τα χέρια όσοι είναι υπέρ. Κατά. Κύριε Άγνιο, παρακαλώ. Ακούσαμε και 189 και 198. Ποια ψηφίζουμε. Γιατί πάμε πολύ γρήγορα στην ψηφοφορία. Θα μπορούσε να είναι η μία ή η άλλη. Ποια είπατε, 189 ή 198. Ποιος είναι υπέρ της 189. Κατά. Διανατάσσεως χειρός είπαμε. Απορρίπτεται. 190 και 191. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπαριθμών 30. Ποιος είναι υπέρ. 30. Έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ή μάλλον καταπίπτει. 194 τώρα. Ποιος είναι υπέρ της 194. Κατά. Απορρίπτεται. 195 τώρα. Ποιος είναι υπέρ της 195. κατά απορρίπτεται 196 ποιος είναι υπέρ της 196 εγκρίνεται τροπολογία 22 ή μάλλον One nine eight. Περνάμε στην 198 τώρα. Ποιο είναι υπέρ. 198. Εγκρίνεται. Εκατόν του κυρίου Δεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Όχι, η 200 έχει καταπέσει. 32. Ποιος είναι υπέρ της 32 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 201. στην υπέρ. Yes. Poprawka Η 200 έχει καταπέσει. 32 εγκρίθηκε. 201 τώρα. Ποιο είναι υπέρ τη 201 της κυρία Κέστιγκερ. Εγκρίνεται. Ο κύριος Τεραμπέλα. Συγγνώμη. Αλλά οι 232 πρέπει να καταπέσουν γιατί εγκρίθηκε 199. Okay, all right. Α, εντάξει. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Οπότε ψηφίζουμε την 33 της ΕΝΒΗ. Όντως πήγαμε πολύ γρήγορα. 33 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Διακόσια του κυρίου Ντεκάστρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Musimy... Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, πρέπει να ψηφίσουμε και τη 202 τη κυρία Χάζκαμπ και του κυρίου Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 202. Κατά. Απορρίπτεται. Τη 203 την ψηφίσαμε. Περνάμε. Στην 200. 205. 205. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 206. Ποιος είναι υπέρ. Έμβη MV34 υπέρ. Εγκρίνεται. 23 της ηγήτριας υπέρ. Εγκρίνεται. 207 του κυρίου Νταντάν. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 208. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 210. 210. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 210. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίθηκε στο παρατρίχα. Πάμε στην τροπολογία 211. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 212. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 233 της κυρία Σράιερ. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογια 2.33 η 38 τη ΕΜΒΗ εγκρίνονται. 220. είναι υπέρ. Για να τάσω στις χειρός παρακαλώ. Εγκρίνεται. 26 της συγκυτρίας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 236, 37 και 38 μαζί τις τρεις τροπολογίες υπέρ εγκρίνονται. 200 239, 239. Ποιος είναι υπέρ. Διανατάσσω της χειρός παρακαλώ. Εγκρίνεται. 240 υπέρ. Ή μάλλον 241 και 242 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Συμβεβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται η συμβαστική 3. Περνάμε στην 246 ε, του κ. Νταντά. Ποιος είναι υπέρ της 246 του κ. Νταντά. Εγκρίνεται. MV40 τώρα. MV40. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 262 και MV42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 263. Σράιερ. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 4. Αλλά προηγουμένως ηλεκτρονικός έλεγχος για την 263. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 263. Τέλος. Απορρίπτεται Λυπάμαι για το λάθος. Αλλά είναι τόσο οριακή η διαφορά. Δεν το πρόσεξα με τα χέρια. Συμβαστική τροπολογία 4 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 271 τώρα. Τσούλο. Ποιος είναι υπέρ της 2.71. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται ψηφοφορία παρακαλώ. Ανοίξτε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 277 του κυρίου Έριξον. Ποιος είναι υπέρ της 277 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 280 του κύριου Νταντά. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 281 ποιος είναι υπέρ ή μάλλον όχι. Α, έχει καταπέσει, συγγνώμη. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 6. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 286. Ποιος είναι υπέρ. Ο διανατάσσεως της χειρός κατά απορρίπτεται 284 και έμβη 45 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτονται 282 και 283 ποιος είναι υπέρ εγκρίνονται Τροπολογία 290. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 32 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Περνάμε στα παραρτήματα. Τροπολογία 291. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 293. 293 είπα. 293. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 294. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 294. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν και κατά τη γνώμη μου έχει απορριφθεί. Ηλεκτρονικά. Ας το ελέγξουμε. Τέλος ψηφοφορία. Ναι, αυτό είχα πει και εγώ. Απορρίπτεται. 295. Ποιος είναι υπέρ. Διανατάσσεω χειρός. 295. Εγκρίνεται. 296. Χάζεκαμπ και εκ. Ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα όμως για την 295. Άρχεται η ψηφοφορία για την 295 του κυρίου Νταντά. Τέλος. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Αυτή τη φορά είχατε δίκιο, κύριε Ταραμπέλα αλλά ήταν οριακή η διαφορά. 296, Χάζενκαπ και ΕΚ. 296, Χάζενκαπ και ΕΚ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμβη 46. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος 46 της έμβη. Κατά. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, τη 46 πάλι, υπέρ, κατά. Απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα. Περνάμε στην τροπολογία 297 του κυρίου Ντεκάστρο και 34 της ηγετρίας. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. 298. Ποιος είναι υπέρ? Διαδικαστικό, κύριος Λαζό. Κύριε Πρόεδρε, στη Γαλλία υπάρχει μια έκφραση που λέει ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, διότι ε, καθώς ψηφίζουμε, εσείς δεν κοιτάτε μπροστά, ε, δεν καταλαβαίνουμε τα ναι, τα όχι. Ε. Ναι, αλλά όταν βλέπω και διαπιστώνω ότι οι τρεις μεγαλύτερες ε, ομάδες είναι υπέρ, βλέπω το ΕΛΚ, τους ε, μεταρρυθμιστές, συντηρητικούς και τους σοσιαλιστές να είναι υπέρ, διαπιστώνω ότι συγκεντρώνουν πλειοψηφία. Αλλά θα κοιτάω και εσάς, εντάξει, θα κοιτάω και εσάς. Πού είμαστε τώρα, πού φτάσαμε. 297 και 34. Ποιος είναι υπέρ. 297 δεκάστρο, 34 σύγκεντρες υπέρ. Εγκρίνονται. 298. Χάζεκαμπ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Έμβη 47. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 47 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 200 ή μάλλον 300. 300 της κυρίας Χάζενκαπ και 48 της ΕΜΒΗ διόρθωση του Πρόεδρου. 301 του κυρίου Τσούλο. Ποιο είναι υπέρ τη 301. Εγκρίνεται. Εμφανώ εγκρίνεται. 305 Νταντά. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 306 της κυρίας Κιώστιγκερ ή όχι. Έμβη 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 309. Ποιος είναι Ηλεκτρονικό έλεγχος όμως πρώτα για την τροπολογία 49 της ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ο κύριος Νταντάν. Κύριε Πρόεδρε, Ξεχάσατε το 305 έχω την εντύπωση κύριε Πρόεδρε. E, Μια στιγμή να το ελέγξουμε επανάληψη της 305. Ποιος είναι υπέρ της 305. Εγκρίνεται. Και ηλεκτρονικός έλεγχος για την 305. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Δαντά. 36 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 36, υπέρ. Υπέρ της 36 της ηγήτριας. Εγκρίνεται. 310 του κυρίου Τσούλο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 311 του κυρίου Ντεκάστρο υπέρ. Εγκρίνεται. 312 και 13. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. 314. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 315 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 και 316. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. 319 και 320. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 319 και 320. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 321. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε μαζί 322 έως 326 όλες μαζί. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών. Εγκρίνονται. 327 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. «3.31» και «MV51». Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία 10. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 343 του κυρίου Αντριέ ποιος είναι υπέρ της 343 και 344 και 345 υπέρ εγκρίνονται. 346 έριξο και 55 Έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη, no vote λέει εδώ, άρα δεν ψηφίζουμε 3.46 και 55. Πάμε στη 42 της κυρίας Χάζεκαμπ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 42. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43 του κυρίου Άγνιου. 43. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. MV3 και 44. όχι, όχι, μόνο την 3 ε, της MV. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 3 της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Κατά. Απορρίπτεται η επανάληψη. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 3 της ΕΜΒΗ. Εγκρίνεται. Ο κύριος Άγνιου. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε στη διερμηνία ε, Μόνο έμβη ακούσαμε, δεν ακούσαμε νούμερο της τροπολογίας. Ποια τροπολογία έμβη ψηφίσαμε, μόνο έμβη άκουσα από την διερμηνία. Έμβη 3 είπα, έμβη 3, τροπολογία 3 της Επιτροπής έμβη, εγκρίνεται... Τροπολογία 44 τώρα. Ή μάλλον 45 και 47 μαζί, 45 και 47 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 46 και έμβη 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 48 και έμβη 5. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 49 τροπολογία. Ερντός. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβεστική ή μάλλον 57. 57 τροπολογία του κυρίου Αρντός. Α, έχει αποσυρθεί. Οπότε πάμε στην ΕΜΒΗ 7. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 7 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58. Νίκολσον Μαγκίνες Γκέρλινγκ Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59, 59 της κυρίας Μίλλερ. Ποιος είναι υπέρ της 59. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 59 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δικό μου λάθος, λέει ο πρόεδρος. 60 της κυρίας Κιώστιγκερ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. 67. Ποιος είναι υπέρ της 67. εγκρίνεται. 68, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 69, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 77, 77 παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ, κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 77. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 81. Ποιος είναι υπέρ. 81. Κατά. Απορρίπτεται. 82 και έμβη 11. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμβη 12 και μια προφορική τροπολογία που την έχετε λάβει. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Έμβη 13. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί, με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση και πάλι το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 73 παράγραφος Β. Ο κύριος Νταντά θέλει το λόγο. Όχι, όχι. Και για τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας όπου προεδρεύει ο εισηγήτρια και απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τους ε, σκιώδεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Απαιτούνται 23 ψήφοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Έχουμε τα δύο τρίτα που απαιτούνται για να είναι έγκυρη για να έγκυρο το αποτέλεσμα, οπότε εγκρίνεται και η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας με πρόεδρο, εισηγήτρια και σκιώδη ηγητές. Συγχαρητήρια κυρία Γιλέρα για την έκθεσή σας και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω θερμά όλους τους σκιώδης ηγητές το τεχνικό επιτελείο, τους βοηθούς. Ε, το θέμα ήταν πολύ τεχνικό, αρκετά δυσνόητο, αλλά μας βοήθησαν όλοι οι εμπειρογνώμονες των ε, πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ θερμά και τη Γραμματεία, τον Κονθάλο, για την αφοσίωση, τη ζέση και την εργότητα προσπάθεια και φυσικά και τη βοηθό μου τη Μαγδαλένα, που θα ήταν αδύνατο χωρίς τη βοήθειά της να τα καταφέρω. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση μπροστά μας και πιστεύω ότι τη μάχη θα την κερδίσουμε. Γιατί θέλουμε να κάμψουμε την μικροβιακή αντοχή, να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών. Αυτό επιδιώκουμε. Στην προηγούμενη ψηφοφορία εγκρίναμε τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα μετά από μια πολύ σημαντική συζήτηση και αυτή η πρόταση θα είναι το επιστέγασμα και μάλιστα στην αρχή, το είδαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ε, η συζήτηση για τον κανονισμό αυτό είναι στενά συνδεδεμένη με τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Γιατί δεν έχει νόημα να ξεκινήσουμε διαπραγμάτευση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές ε, μετά τα κτηνιατρικά φάρμακα. Θα γίνουν εκ παραλίλου λοιπόν και με τις σκιώδεις ηγητές θα εξασφαλίσουμε ένα συντονισμό των εργασιών με την Επιτροπή ΕΜΒΗ, με την κυρία Γκροστέτ που είναι συγκήτρια για τα κτηνιατρικά φάρμακα, για να αποφύγουμε στρεβλώσεις ή αντιφάσεις μεταξύ των δύο κανονισμών, που επαναλαμβάνω πρέπει να δρομολογηθούν εκ παραλλήλου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αγγιλέρα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τα συμφέροντα των γεωργών. Γιατί το πρόβλημα είναι δύσκολο, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όμως να κρατήσουμε μια ισορροπία στο τέλος μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων. να μην ξεχνούμε και τους ε, γεωργούς και τους παραγωγούς μας. Και φυσικά την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, ε, της ευρωπαϊκής αγοράς σε σχέση με τις αγορές τρίτων χωρών. Πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια, τους σκιώδεις εισηγητές, ε, τους συνεργάτες και βοηθούς και περνάμε στο σημείο 8. Τη βελτίωση της καινοτομία και τη οικονομική ανάπτυξη στη διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντο. Επίση σημαντικό θέμα. να μην κάνω εγώ την εισαγωγή, καλύτερα να την αφήσω στον εισηγητή μας, τον κύριο Χαϊτεμα. Παρακαλώ. <clears throat> Eh, ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι πάρα πολύ που δημιουργώ ε, τέτοια προβλήματα. Θα ήθελα να ζητήσω όμως από την Επιτροπή να αναβάλει την ψηφοφορία και το πρόβλημα είναι ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Όσον αφορά ε, το περιεχόμενο είναι εντάξει, αλλά στα συν πλην δυστυχώς ε, κάποια σημεία είναι παραπλανητικά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή που επέστησε την προσοχή μου στο θέμα αυτό. Για να είμαστε όμως κατά 100% σίγουροι ότι δεν θα γίνει κανένα λάθος, θα θέλαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Δεν βλέπω παρατηρήσεις από τους συναδέλφους. Οπότε και η γραμματεία δεν έχει σχόλια και άρα δεχόμαστε την πρόταση του εισηγητού και αναβάλουμε την ψηφοφορία της έκθεσης γιατί είναι σημαντικό για τόσο σημαντικό θέμα να καταλήξουμε σε συμφωνία. Γι' αυτό και συμφωνούμε με τη σύσταση του εισηγητού και αναβάλουμε την ψηφοφορία της έκθεσης Χαϊτεμα. Περνάμε στο επόμενο λεπτό θέμα. Την ε, γνωμοδότηση της κυρίας Σκοτ Κάτω, τη νέα συμμαχία, μάλλον ο πρόεδρος ε, μιλάει για τη έκθεση Μπόγκοβιτς που είναι για συζήτηση, την έκθεση πρόοδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ξέχασα λέει ο πρόεδρος ε, μία ψηφοφορία ακόμη την ψηφοφορία για την γνωμοδότηση με θέμα τη Νέα Συμμαχία για την Επισητιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή. Αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης. Η δική μας Επιτροπή εκπόνησης γνωμοδότηση με συντάκτρια την κυρία Μόλι Σκότ Κάτω από τους Πράσινους. Έχουμε 152 τροπολογίες αλλά και κάποιες συμβιβαστικές για, την οποία για τις οποίες ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Και δεν ξέρω αν θέλει το λόγο η κυρία Σκοτ κάτω πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όχι, οπότε περνάμε στην ψηφοφορία της γνωμοδότησης, των τροπολογιών πρώτα. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της και πάλι. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ε, Ποιο είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε κατευθείαν στη συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και η συμβαστική τροπολογία 2. Περνάμε στην τροπολογία 24 της κυρίας Νόεχλ. 24 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 24 της κυρίας Νόεχλ, άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 27. Ποιος είναι υπέρ της 27. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Και περνάμε στην τροπολογία 45. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Είναι της κυρίας Κάτω της ηγετρίας υπέρ. Εγκρίνεται η 45. Συμβαστική τροπολογία 4. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας για τη συμβαστική τροπολογία 5. Περνάμε στην 63 τώρα. Βιέγκας και Σένερα. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται η 63. Περνάμε στη συμβαστική 6, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 122 λέει ο πρόεδρος. Ταραμπέλη και Νόιχλ. Ποιο είναι υπέρ. 122. Εγκρίνεται 122 Μπράνεν, Ταραμπέλα και Νόιχλ. Περνάμε στην 102 της εισηγήτριας Σκοτ Κάτω. Ποιος είναι υπέρ της 102. Εγκρίνεται και αυτή. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. Τέλος. Εγκρίνεται. 148 τροπολογία. Μπράνεν, Ταραμπέλα και Νόιχλ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 149. Εκ, Χάζενκαπ, Βιέγκας και Σένρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. 150 της κυρίας Νόιχλ. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 150 Νόιχλ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Ε, οριακά πέρασε. Ε, μάλλον απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Απορρίπτεται 150. Πάμε στην 151. Ριμπέιρο. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Και 152 της κυρίας Ριμπέιρο. Υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης με τις τροπολογίες. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια και την συντάκτρια γνωμοδότηση, συντάκτρια γνωμοδότησης για την εκπόνηση ε, και της γνωμοδότησης και των συμβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστούμε και τέτοιες γνωμοδοτήσεις χρειαζόμαστε. Περνάμε στο σημείο 10 τώρα. α, συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί χθε σας υποσχέθηκα δύο πράγματα. Πρώτον, προσοχή παρακαλώ. Μια πολύ σημαντική πληροφορία να σας δώσω. Χθες υποσχέθηκα ότι ένα σημείο θα το αναβάλουμε για σήμερα αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Την ενημέρωση που θα μας κάνει ο κύριος Χόισλινγκ για την πρόοδο των εργασιών στις διαπραγματεύσεις ε, του τριμερούς διαλόγου. Θα θέλατε κυρία Χόισλινγκ να μας κάνετε τώρα την ενημέρωση. Σας δίνω λίγα λεπτά να προετοιμαστείτε και να σας ε, δώσω μια άλλη πληροφορία. Καταρχήν έστειλα επιστολή στον πρόεδρο Γιουνκέρ επισημένοντας την έκτακτη κατάσταση και τα προβλήματα εξαιτίας της κρίσης στις γεωργικές αγορές, στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Γιατί στο Παρίσι συναντήθηκα με πολλούς γεωργούς και επηρεάστηκα από τη θέση τους και είχαμε και την έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα στη συνάντηση με τον Επίτροπο Χόγκαν για τα προβλήματα αυτά και την κρίση στην αγορά των γεωρικών προϊόντων. Ζήτησε λοιπόν μια παρέμβαση στην αγορά γεωργικών προϊόντων. Σας έστειλα αντίγραφο τη επιστολή που έστειλα στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον πρόεδρο Γιούγκερ. Και επίση θα πρέπει να ενισχυθούν και οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του αρμοδίου επιτρόπου, του κυρίου Χόγκαν. Γιατί έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος του 2015 κάποιες προσπάθειες προώθηση και ανέβρεση νέων αγορών ε, για τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την έκτακτη κρίση που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Είχαμε, επαναλαμβάνω, τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας όπου επισημάνουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο κύριος Νίκολσον. Yes, chairman. Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ που ήρθατε σε επαφή με τον Επίτροπο για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει όμως να πω ότι είμαι λιγότερο ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την Επιτροπή. Ο Επίτροπος την προηγούμενη Δευτέρα μας επισκέφθηκε στο Στρασβούργο επί μια μισή ώρα. Όλοι είχαμε να του πούμε τα παράπονά μας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί σε όλη την Ευρώπη δεν είναι προβλήματα γεωργών σε μια περιφέρεια ή σε μια χώρα, είναι προβλήματα γεωργών παντού. Μιλήσαμε για τον γαλακτοκομικό τομέα, τον χειροτροφικό, τον, ε, τομέα του βοηού κρέατος. Ε, και λόγια, λόγια, λόγια, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Θέλω ε, ο Επίτροπος να έρθει στην Επιτροπή μας μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου και να μας πει τι θα κάνει. Όχι να μας διαβάζει ανακοινοθέντα τύπου. Είπατε και εσείς, ε, όλοι μας συναντιόμαστε με ε, γεωργούς ε, στις εκλογικές μας περιφέρειες. Μερικοί θα μείνουν από δουλειά και είδαμε και στο Στρασβούργο τη συνάντηση όπου ακούσαμε ότι αυτοκτονούν οι Γεωργοί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο δομημένη προσέγγιση και δεν έχει νόημα απλά να συνεχίσουμε να μιλάμε. Οι Γεωργοί περιμένουν πράξεις, όχι λόγια μόνο. Και κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σε επαφή με τον Επίτροπο και χαίρομαι που ο Επίτροπος παραδέχεται ότι αντιμετωπίζουμε κρίση, αλλά η κρίση αφορά ε, το σύνολο του γεωργικού τομέα και όχι μόνο τον γαλακτοκομικό. Εάν δεν ενεργήσουμε γρήγορα και αν δεν ε, παρουσιάσουμε εδώ τις απόψεις τους, ε, τότε θα χάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο. Επαναλαμβάνω, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους, ε, στη διάσκεψη ε, Προέδρων Επιτροπών, στη συνάντηση που είχαμε με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν, επίση επισήμανα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μα και την κρίση που διανύει ο κλάδο. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσει. Χθε ο Επίτροπο Χόμπεν, ε, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Οργίας. Από ό,τι ξέρω έγινε συζήτηση, αλλά δεν είναι οριστική απόφαση. Γιατί αναφέρθηκε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προετοιμασίες. Γιατί αυτό περιμένουν οι υπουργοί, συγκεκριμένες προτάσεις δεν υπήρχε μεγάλη διάσταση απόψεων. Υπήρχε μάλλον ε, θετική ανταπόκριση την ε, πρόταση του Υπουργού Γεωργίας της Γαλλίας. Αυτά λένε οι δικές μου πληροφορίες. Αλλά περιμένουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από τα συμπεράσματα του χθεσινού Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας. Για να τα μοιράσουμε στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Κατόπιν ε, θα, θα ακολουθήσουν γραπτές διαβουλεύσεις ε, με συνοπτικές διαδικασίες για να μην περιμένουμε ε, την επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον. Γιατί γνωρίζουμε πόσο δεν είναι η κατάσταση. Είχαμε πολύ συναντήσεις με εκπροσώπους του κλάδου και στη Γαλλία και στην Πολωνία και ακριβώς εμείς τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας που περισσότεροι είμαστε και γεωργοί έχουμε άμεση επαφή με τους ε, γεωργούς και ξέρουμε την κατάσταση που περνάνε. Μία σύντομη παρακαλώ ανταλλαγή απόψεων γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο για εκτένη συζήτηση. Ο κύριος Άγνιου πρώτα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για να συζητήσουμε για το χθεσινό Συμβούλιο Γεωργίας, όπου όπως φαίνεται, παρότι περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις, ότι έγιναν κάποιες προτάσεις ε, βάσει των όσων συζητήσαμε με τον κύριο Επίτροπο. Αυτό που εμένα μου δημιουργεί ερωτηματικά για τη διαδικασία είναι το πόσο αργά κινούνται τα πράγματα. Είχαμε πει στον Επίτροπο εμείς εδώ και δύο χρόνια ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, διότι είμαστε σε άμεση επαφή με πολλούς επαγγελματίες και αυτό που μου δημιουργεί ερωτηματικά είναι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που ελήφθησαν χθε ε, πώς βλέπει τη δική μας συνέλευση ο Επίτροπος. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων Γεωργών, είμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους και όταν μας λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε όλα τα κράτη-μέλη, πιστεύω ότι επιβάλλεται να εισακουστούν, να μας ακούσει ο κύριος Επίτροπος, ε, όχι να έρχεται μπροστά μας και να μας λέει το σκέφτομαι. Την περασμένη εβδομάδα, όταν στο Στρασβούργο, ε, ελπίζαμε να ακούσουμε προτάσεις από αυτόν ε, τις οποίες τα υπέβαλε στο χθεσινό Συμβουλίο Γεωργίας. Αυτό εμένα μου δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά το δημοκρατικό μας ρόλο και το ρόλο που παίζει η Κομισιόν. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Ενστανιζόμαστε τις απόψεις σας. Ας μην επαναλαμβανόμαστε. Τη Δευτέρα ο Επίτροπος Χόγκαν ε, ήθελε ε, πρώτα να υποβάλει επισήμω τις προτάσεις στους υπουργού και μετά σε εμά. Χθε το έκανε. Δεν γνωρίζουμε τις ε, λεπτομέρειες, θα μάθουμε και τις λεπτομέρειες, τότε θα λάβουμε απόφαση. Παρακαλώ να είστε σύντομοι παρεμβάσει. παρεμβάσεις, να μην γίνει εκτενή συζήτηση, δεν υπάρχει χρόνος. Ο κύριος Άγνιου δεν θέλει το λόγο, οπότε ο κύριο Χόισλινγκ ή μήπω δεν θέλει. Όχι, ο κύριο Χόισλινγκ ich stimme voll Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Νίκολσον. Δεν μπορούμε να θεσπίσουμε κανόνα ε, να έρχεται ο Επίτροπος ε, Γεωργίας ε, κάθε φορά μετά από Υπουργικό Συμβούλιο. Διότι εγώ προβληματίζομαι που τόσο σπάνια βλέπουμε τον Επίτροπο, ε, διότι έχει τόσα πολλά ταξίδια. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κύριο Σταραμπέλα. Πριν από ακριβώ ένα χρόνο, εγώ είχα ανακοινώσει αυτή την κρίση στη χώρα μου γιατί ήταν αναπόφευκτη. Αλλά εμεί τη δημιουργήσαμε. Αυτή τη στιγμή εγκαταλείπουμε ε, ο ένας μετά τον άλλο τους μηχανισμούς ρύθμισης παραγωγής. Ε, ε, αυτό δείχνει τι συμβαίνει. Δεν έχουμε κανένα μηχανισμό ασφάλειας αποτελεσματικό όσον αφορά το γάλα. Αντίθετα από τις Ηνωμένες όπου βοηθούν τους παραγωγούς ανεξάρτητα από τις εξελίξεις της αγοράς. Τώρα στην παγκόσμια αγορά οι τιμές ε, χαμηλώνουν και διαπραγματευόμαστε και συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί τη γεωργία μεγάλη προτεραιότητα. Είναι το τελευταίο πράγμα που διαπραγματεύεται. Θα πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν πώς λειτουργούμε, πώς χρηματοδοτούμε την γεωργία. Έχει ήδη πεθάνει σήμερα η γεωργική πολιτική, ενώ θα έπρεπε να υποστηρίζει τους γεωργού. Αυτό ήταν, αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός της πολιτική. Ε, πολιτικής, να υπάρχει ποιότητα, καλέ τιμέ, ε, να εξασφαλίζει εισόδημα στους γεωργού. Έχουμε αποτύχει σε όλα αυτά. Οπότε πρέπει να δούμε το συντομότερο δυνατόν τι θα γίνει με την κοινή γεωργική πολιτική, όχι σε πέντε χρόνια, ε, για να δούμε πώ θα δημιουργήσουμε μηχανισμού για να βοηθήσουμε του γεωργού. Αλλά κάποια στιγμή, για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να ελέγχουμε την παραγωγή. Αν την αφήσουμε ελεύθερη, θα επιστρέψουμε στη δεκαετία του 80, όπου τα πράγματα θα είναι πολύ ακριβά ε, ή θα ε, έχουμε ανθρώπου που θα καταστρέφουν τα τρόφιμα και θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό που να αντιστοιχεί η προσφορά στη ζήτηση. Μα συμφωνώ Αυτά να το πείτε όμως στον Επίτροπο. Γιατί με τον Επίτροπο όλοι είμαστε ευγενικοί, συμπαθητικοί. Μα γι' αυτό είχαμε τη συνάντηση με τον Επίτροπο για να τα πούμε κατά πρόσωπο, έξω από τα δόντια. Έπρεπε να φανεί αυτή η γενικευμένη δυσαρέσκεια στην Επιτροπή. Παρακαλώ, ένα λεπτό καθένας, όχι παραπάνω, γιατί αυτό ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Σένερα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ να έρθει ο Επιτρόπος και να μας εξηγήσει τι συμφώνησαν ε, χθες οι Υπουργοί Γεωργίας, αν συμφώνησαν κάτι τελικά. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής μείωσης ε, των κτηνοτρόφων. Πώς θα γίνει όμως κάτι τέτοιο. Θα είναι ένας νέος τρόπος για να αποπέμψουμε από τον κλάδο τους ε, μικρής εμβέλειας κτηνοτρόφους, γιατί είναι και αυτό πιθανό. Γιατί είδαμε και άλλες ε, στηρίξεις οικειοθελούς εγκατάλειψης της παραγωγής. Αλλά αυτοί που εγκατέλειπαν την παραγωγή κυρίω ήταν οι μικροκαλλιεργητές. Θα το κάνουμε και με τους κτηνοτρόφους και με ποιο τρόπο. Επίσης, διαρωτώ με και ρωτώ και εσάς, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας θα ταχθούν υπέρ της ρύθμισης της ε, παραγωγής και θα απαιτήσουμε ρύθμιση της παραγωγής. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουμε την κρίση κατά τη γνώμη με ρύθμιση της παραγωγής. Ο κύριος Ροπέ, ένα λεπτό παρακαλώ μόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που θίξατε το θέμα αυτό. Χαίρομαι που συναντήσατε συνάντηση με τον Επίτροπο στο Στρασβούρο και που στείλατε επιστολή στον κύριο Γιούνκερ. Ναι, πιστεύω και εγώ ότι μας αξίζει μια απάντηση. Ο Επίτροπος υποσχέθηκε εντός μιας εβδομάδας να θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό της προσφοράς στην αγορά η προθεσμία έληξε χθε και δεν έχουμε δει ακόμα προτάσεις στο Συμβούλιο. Από ό,τι γνωρίζω, είπε ότι θα χρειαστούν τρει μήνες για να αναλύσουν την κατάσταση της αγοράς και τότε θα υποβάλουν προτάσεις. Νομίζω ότι παιχνίδια παίζει. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος ε, θα έπρεπε να έρθει εδώ και να μας ε, εξηγήσει την κατάσταση. Οι γεωργοί σε όλες τις χώρες ε, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Συνομίλησα με Γεωργού στη χώρα μου και του είπα ότι στο Στρασβούργο θα δούμε πλήρη πρόταση και τίποτα δεν είδαμε. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι μέλος της Επιτροπής ε, αυτής εδώ και πολύ καιρό και χθες πήγα στην ιστοσελίδα για να ψάξω να βρω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και πρέπει να πω ότι ο Επίτροπος ε, σε σχέση με τις παρεμβάσεις με το όριο των παρεμβάσεων ανέφερε κάτι και αναφέρει ότι μπορεί τον Απρίλιο να έχουμε περαιτέρω μείωση των τιμών καθώς θα αρχίσουμε να φτάνουμε στους όγκους που ε, συζητήθηκε. Αυτό που προτείνει όμως είναι ε, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα μέτρα, αλλά βραχυπρόθεσμα αποκλείεται να αποφύγουμε την κρίση που εποάζεται. Όσον αφορά την εθελοντική ε, διαχείριση, είναι ένα προσωρινό μέτρο και όσον αφορά τι αυξήσει παραγωγή στα κράτη-μέλη, ελάχιστα θα κάνουμε για να επηρεάσουμε τι αγορέ. Χρειαζόμαστε περαιτέρω άμεσα μέτρα, πιστεύω. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, όταν κάποιος ε, κάνει αίτηση για δουλειά, εξετάζουμε το βιογραφικό του. Είναι λοιπόν ε, περίεργο που τα Ιρλανδικά μέλη του Κοινοβουλίου διαφωνούν με τον Ιρλανδό Επίτροπο. Αλλά δεν διαφωνούμε με τον Ιρλανδό Επίτροπο, διαφωνούμε συγκεκριμένα με τον κύριο Φιλ Χόγκαν. Ε, θα έπρεπε να είχατε διαβάσει το βιογραφικό του, ε, θα έπρεπε να μας είχατε ακούσει τότε πριν ε, τον ορίσετε Επίτροπο. Δεν νομίζω ότι είστε στο θέμα μας. Και τέτοιες παρεμβάσεις δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δεν θα ήθελα να μεταφέρετε εδώ τοπικέ χώρε συζητήσει, εθνικέ στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε, έτσι φαίνεται να έχετε πολύ συναρπαστική η συζήτηση με αυτόν τον τρόπο και η ελευθερία λόγου φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να πω ότι εγώ εξέτασα τις χθεσινές εκθέσεις και είδα και εννέα μέτρα να προτείνονται ορισμένα έχουν υιοθετηθεί, αλλά δεν είναι σαφές το πόσο αποτελεσματικά θα είναι. Θα μας βοηθούσε να ήταν εδώ ο Επιτροπός σήμερα το πρωί. Πρέπει να δούμε λοιπόν κατά πόσο υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά η συζήτηση είναι ευρύτερη. Ορισμένοι λένε ότι αν ελέγξουμε την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωθούν οι τιμέ. Αλλά μακάρι να ήταν έτσι ο κόσμο σήμερα, αλλά δυστυχώ δεν είναι. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια συζήτηση για του μελλοντικού προσανατολισμού τη κοινή γεωργική πολιτική πέραν της απόκρισης στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να ξανακαλέσουμε εδώ τον Επίτροπο για να μας εξηγήσει τα εννέα αυτά μέτρα τι θα επηρεάσουν, ποιο θα τα χρηματοδοτήσει. Υπάρχουν αρκετά λεφτά στον προπολογισμό. Το μεγάλο ερώτημα για τον Γιούνκερ είναι ότι αυτή τη στιγμή οι γεωργοί ε, πληρώνουν το πολιτικό κόστος ε, ε, του εμπάργου της Ρωσίας και θα πρέπει να μας εξηγήσει τι γίνεται με όλο αυτό. Θα πρέπει να έρθει εδώ στην Επιτροπή μα και να μας ακούσει. Αυτό το ανέφερα στην επιστολή. Ότι θα πρέπει ε, να ε, φροντίσουμε ώστε να αρθεί το ρωσικό εμπάργο γιατί ε, είναι τεράστιο το κόστος για τους γεωργούς που ανέλαβαν να πληρώσουν τα σπασμένα του εμπάργου. Και μάλιστα το, τη Δευτέρα στις 4, ε, παρουσία του Επιτρόπου Χάν που είναι αρμόδιος, ανέφερθηκε η ανάγκη ε, άρσης του ρωσικού εμπάργου. Ε, το επισήμανε και μάλιστα πολύ έντονα. Πρέπει επιτέλους να αρθεί το ρωσικό εμπάργο γιατί ε, υφίσταται τα πάντα εξαιτία του Γιώργη. Πάντως ε, έχουμε χρόνο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση για να λάβουμε τις πληροφορίες από τον Επίτροπο και να ενημερωθούμε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας. Αλλά λεπτομέρειες, όχι απλώς γενικές και αόριστες ε, δηλώσεις για τα συμπεράσματα. Γιατί αυτό ζήτησαν και οι Υπουργοί, να συγκεκριμενοποιηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιτρόπου Χόγκαν. Και αυτό θέλουμε και εμείς να μάθουμε τις λεπτομέρειες και ε, συνήθως δεν θέλει εκ των προτέρων να παρουσιάζει τι ε, προτάσει ο Επίτροπο Χόγκαν πριν τις παρουσιάσει επίσημα στους υπουργούς. Γιατί στις 7 του μηνό που είχαμε τη συνάντηση είπε ότι δεν θέλει να πει τις λεπτομέρειες γιατί αμέσως ε, θα διατυπωθούν ε, επιπλέον απαιτήσει και γι' αυτό προτίμησε πρώτα να περιμένει το Συμβούλιο Υπουργών. Αυτά κλείνει προς το παρόν η συζήτηση. Ο κύριος Δαντά, αλλά όχι άλλος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ όπως και όλοι οι υπόλοιποι συναδέλφοι έλαβα γνώση των προτάσεων που έγιναν χθε. Αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι όλα αυτά δεν χρηματοδοτούνται. Και εκεί τίθεται το εξή ερώτημα, το οποίο είχα αναφέρει και εγώ όταν συζητήσαμε την ενιαία οργάνωση τη αγορά την οργάνωση τη ενιαία αγορά, ότι όταν παρεμβαίνουμε με εργαλεία αντιμετώπιση τη ε, κρίση, παίρνουμε λεφτά από τι πιστώσει που θα έπρεπε να δώσουμε από τον πρώτο πυλώνα στου γεωργού το επόμενο έτο. Δηλαδή, του ε, επιβάλλουμε δύο πρόστιμα. Μία φορά τη στιγμή της κρίσης διότι τα επίπεδα αρρωγής μας δεν μπορούν να καλύψουν απόλυτα να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης και τους ε, επιβάλλουμε και άλλο πρόστιμο το επόμενο έτος γιατί δεν λαμβάνουν το επίπεδο αρρωγής του πρώτου πυλώνα που κανονικά δικαιούνται. Πιστεύω λοιπόν ότι δεδομένη τώρα τη κρίση και των αιτιών τη και του ζητήματο του εμπάργου στο οποίο πρέπει να διτεθούμε πρέπει να στραφούμε στον κύριο Γιούνκερ ώστε να λάβουμε χρηματοδοτικά κονδύλια για να καλυφθούν ε, τα προβλήματα αυτά. Αλλά ενδεχομένω να υπάρχουν τέτοια κονδύλια που να μπορούν να ανταποκριθούν, να, να μα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική και τη γεωργική κρίση ταυτόχρονα. Αν αυξήσουμε διατροφικά κονδύλια, θα δώσουμε περισσότερα λεφτά στους γεωργούς και θα θρέψουμε και τους μετανάστες. Αυτό κάνουν και οι Αμερικανοί. Καλό θα ήταν μια, μια φορά να εμπνευστούμε από τις ΗΠΑ ενδεχομένω. Ναι. Αυτό επισημάναμε και στον Επίτροπο Χάν τη Δευτέρα στις 4. Θέλετε τίποτα καινούριο να προσθέσετε, κύριε Μπούντα. Πολύ σύντομα παρακαλώ, δύο λόγια. Πολύ πολύ σύντομα, επιγραμματικά. Ε, δύο λόγια κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν έχουμε υπερβολική παραγωγή είτε γάλακτος είτε χειριοκρέατος χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στην αγορά για να δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς για να επαναπροσανατολιστούν σε άλλες καλλιέργειες και σε άλλη ε, ειδικτυνοτροφία, τα προβλήματα θα πολλαπλασιάζονται είναι αναπόφευκτο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια γρήγορη λύση. Ευχαριστώ. Σα συγκετεύω. Α μην επαναλαμβάνουμε πράγματα που ήδη υπόθηκαν. Ο κύριο Σελιμόβιτς. Ναι, ευχαριστώ. Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο σα, αλλά να πω το εξή Τα συζητήσαμε, το συζητήσαμε αυτό το ζήτημα, τα διάφορα προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση και υπόθηκε σαφέστατα ότι το εμπάργκο είναι μόνο ένα από τα προβλήματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ορισμένε χώρε και καθόλου πρόβλημα για άλλε χώρε, διότι δεν είχαν εκτεθεί καθόλου στη Ρωσία. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια πλήρη εικόνα όλων των αιτιών που οδηγούν στην κρίση και ορισμένα μέτρα αντιμετώπιση του. Διότι η κρίση αυτή είναι μεγάλη και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα των προβλημάτων που οδηγούν στην κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φλάναγκαν, και εσεί παρακαλώ, επιγραμματικά και εντό θέματο, όχι εκτό θέματο. Θα είμαι σύντομο. Η αλήθεια πονάει. Θα παραμείνω στο θέμα, αλλά η αλήθεια πονάει. Ναι. Ε, φυσικά πονάει η αλήθεια και σε άλλους πονάει γιατί έχουν πρόβλημα υγείας. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα στείλουμε επιστολή στον Επίτροπο Χόγκαν. Αλλά παρακαλώ τα ίδια να τα πείτε και στις πολιτικές ομάδες σας. Για να φτάσει και στη διάσκεψη των Προέδρων. Όχι ε, την ε, πέμπτη στις τέσσερις ε, τελευταία στιγμή να βγαίνει αυτό το θέμα. Και ήταν παρόν ο Επίτροπος Χάν και ευχαριστώ όσους ε, ήταν από τις πολιτικές ομάδες γιατί ήταν τέσσερις το απόγευμα πέμπτη Πέμπτη, 4 το απόγευμα και παρόλα αυτά καταφέραμε να παρουσιάσουμε καλά το θέμα στον Επίτροπο Χάν. Και περνάμε τώρα στην ενημέρωση από τον κύριο Χόισλινγκ. Πάντως να έχετε υπόψη ότι και το δικό σας θέμα αναφέρθηκε εκεί. Πρόεδρε, απλά θα ήθελα να διορθώσω κάτι. Είπατε ότι όλοι ήταν ευγενικοί απέναντι στον Επίτροπο την προηγούμενη φορά. Δεν θα συμφωνήσω. Όσον αφορά τον τριμερή διάλογο, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ε, συνάντηση όπου συζητήθηκε το εμπόριο. και οι κανόνες παραγωγής ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το θέμα των εισαγωγών. Και τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι το παρόν σύστημα με την ευέλικτη ισοδυναμία δεν αρκεί και η Κομισιόν πρότεινε για τις εισαγωγές να ισχύει η συμμόρφωση. Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ καλό, αλλά στην πράξη είναι σχετικά δύσκολο διότι αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν κατά 100% τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάτι που είναι αδύνατον. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες ε, κατά τις εισαγωγές. Για το Κοινοβούλιο ήταν σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές ε, συνθήκες και περιβαλλοντικά θέματα κατά τις εισαγωγές. Ε, καταλήξαμε σε συμβιβασμό ανάμεσα στη θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά σε ένα θέμα δεν συμφωνούμε, το οποίο ε, διέπει το σύνολο των διαπραγματεύσεων. προκύπτει συνεχώς το θέμα των κατεξουδότηση των εκτελεστικών πράξεων. Ε, το Κοινοβούλιο ε, δεν μπορεί να δεχτεί να ισχύουν αποκλειστικά οι κατεξουδότηση πράξης. Ε, έχουμε αναβάλει λίγο το θέμα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε τελικά απόφαση. Και είχαμε και το θέμα των μεικτών εκμεταλλεύσεων. μπορούμε να τις δεχτούμε μόνο εάν οι διάφορες παραγωγές είναι αυστηρά διαχωρισμένες. Και ζητήθηκε στα ψάρια να μην ισχύει αυτό. Το Κοινοβούλιο, σε ενόηση με τον ε, αρμόδιο εισηγητή, ε, είπε ότι δεν μπορούμε να μην έχουμε διάκριση και στα ψάρια, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ε, ανακατεμένα τα βιολογικά με τα, τους βιολογικούς με τους μη βιολογικούς σολομούς. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε τους ε, κανόνες εφαρμογής, ε, διότι στους κανόνες ε, της Επιτροπής ε, δεν προβλεπόντουσαν αυτές οι περιπτώσεις, σε περίπτωση που συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο σε κάποια σημαντικά σημεία. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη. Προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε πάνω στα σημαντικά θέματα. Τώρα το αν τελικά θα έχουμε ε, επιτυχία αυτό θα φανεί. Ε, τίθεται το θέμα πάντα των ε, κατοξιδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Ε, ελπίζουμε να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε γρήγορα στο θέμα αυτό. Αλλά ε, πάντα στη διαπραγματεύση με το, κοινο, Συμβούλιο έχουμε το πρόβλημα ότι πεισματώνει το Συμβούλιο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι το κλίμα ήταν αρκετά καλό και στον τελευταίο και στους προηγούμενους τριμερείς διαλόγους και πιστεύω ότι κατά την επόμενη συνάντηση θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε χωρίς να απεμπολίσουμε τα αιτήματά μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε λακωνικοί, ε, κύριοι Νίκολσον και Ταραμπέλα. Παρακαλώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Νίκολσον. Ο κύριος Νίκολσον, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για ε, τις παρατηρήσεις του. Στην πατρίδα μου είχα πρόσφατα συνάντηση με μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται ε, με τις βιολογικές μικτές, σύνθετες ζωοτροφές. στην ε, Βόρεια Ιρλανδία αλλά ε, και στην νήσο της Βρετανίας έχουν μεγάλη εγκατάσταση. Συζητήσαμε λοιπόν από πού προέρχονται οι πρώτες ύλες τους. ασχολούνται και με την ε, έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά ε, το θέμα των ζωοτροφών και την βιωσιμότητα του τομέα. Υπάρχουν ανησυχίες ε, σχετικά με τις επιπτώσεις των τροπολογιών στο σύνολο του τομέα αυτού, ιδιαίτερα την χειροτροφία και τα πουλερικά. διότι υπάρχουν ανεπαρκείς εισαγόμενες ζωοτροφές καθώς και ε, εγχώρια παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα Απαιτείται λοιπόν το 30% να παράγεται σε συνεργασία με βιολογικές εκμεταλλεύσεις, ε, κάτι που στην πράξη θα είναι απολύτως ανέφικτο στον πραγματικό κόσμο. Με ανησυχεί το θέμα αυτό, διότι αν ακολουθήσουμε την οδό αυτή, και θα χαρώ αν ο εισηγητής μου πει ότι όχι δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την οδό, διότι διαφέρει κιόλα η ερμηνεία των διαφόρων οδηγιών στις διάφορες περιφέρειες. Ε, χρειαζόμαστε όμως επανεξέταση της ε, αγοράς βιολογικών ζωοτροφών. Είναι όμως εκπληκτικό το πώς αναπτύσσεται ο τομέας αυτός ε, και δεν έχουμε επαρκείς πρώτες ύλες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν οι καταναλωτές το θέλουν, οι παραγωγοί το θέλουν, αλλά δεν υπάρχουν οι πρώτες ύλες και εξαρτόμαστε από εισαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς και όλας καμία εγγύηση ότι πληρούν τα πρότυπα οι ζωοτροφές αυτές, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση στην αγορά ζωοτροφών. Ελπίζω μάλιστα να μην δημιουργούμε περισσότερη γραφειοκρατία. Είναι ένα θέμα που ανησυχεί πολλούς, η καλλιέργεια δηλαδή βιολογικών ζωοτροφών. Οι άνθρωποι που ασχολούνται στον τομέα αυτών ενδιαφέρονται πολύ για το θέμα και θέλουν την ανάπτυξη του τομέα. Αλλά θα πρέπει να ακούσουμε τις ανησυχίες τους και ελπίζω ως εισηγητής να μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Έχουμε πρόβλημα με το χρόνο τώρα. Το καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε. Κύριο Σταραμπέλα. Υπόσχομαι, Πρόεδρε, μόνο για δύο λεπτά θα μιλήσω. Ο βιολογικός τομέας φυσικά επεκτείνεται διαρκώς ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιστοιχεί σήμερα σε 22 δισεκατομμύρια ευρώ συναλλαγών πανευρωπαϊκά. Και δεν έχουμε αρκετούς παραγωγούς στην Ευρώπη. Ε, έτσι έχουμε λοιπόν μαζικές εισαγωγές, οπότε πρέπει να είμαστε ε, πολύ αποφασιστικοί εκεί. Η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να απαιτήσει πολύ αυστηρούς κανόνες για τις εισαγωγές. Δεν μπορούμε να εισάγουμε οτιδήποτε χωρίς ελέγχους. Ε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους ελέγχους, διότι αλλιώς μπορεί να υπάρξει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με ψευδείς επιγραφές βιολογικής παραγωγής και να δημιουργηθεί αθέμητος ανταγωνισμός για τους ευρωπαϊκούς παραγωγούς. Δεύτερον, οι μεικτές εκμεταλλεύσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ διότι η βιολογική παραγωγή είναι κάτι στο οποίο πρέπει να πιστεύουμε, ε, να χρησιμοποιούμε αυτές τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ε, ε, μέσω μεθόδων να εγκαταλείψουν συγγνώμη τις παραδοσιακές μεθόδους χρησιμοποιώντας μεθόδους καλλιέργειας χωρίς χημικά ναι, είναι μία τάση σήμερα η βιολογική παραγωγή. Ναι, θα μπορούσαμε να δεχθούμε τη μεικτή παραγωγή, αλλά σε μια εκμετάλλευση που θέλει να ε, διαφοροποιήσει ένα κομμάτι της παραγωγής με βιολογική παραγωγή ε, θα πρέπει ας πούμε αν ε, παράγει πουλερικά βιολογικής παραγωγής να χρησιμοποιεί βιολογικά τρόφιμα, βιολογικές ζωοτροφές από την ίδια γεωργία. εάν δεν τα εφαρμόσουμε αυτά, ξέρω ότι η Ιταλία και το Βέλγιο τα εφαρμόζουν, αλλιώς οι βιολογικές, ε, οι βιολογικές, τα βιολογικά τρόφιμα θα μολυνθούν, θα επιμολυνθούν από μη βιολογικές παραγωγές. Εδώ εκπροσωπώ εγώ τους μικρούς παραγωγούς οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οι οποίοι δεν έχουν φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς και τους βιολογικούς παραγωγούς. Σας ευχαριστώ που δείχνετε κατανόηση για το πρόβλημα με το χρόνο που έχουμε. Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι λακωνικός. Λίγα σχόλια έχω μόνο. Καταρχήν ευχαριστήσω το συνάδελφο Μάρτιν Χόισλινγκ για το πολύ καλό το έγγραφο σας εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω να πετύχετε τους στόχους σας. Σε ό,τι αφορά τις μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μερικέ, μερικά κρατημέρια έχουν τέτοιες μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις με βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες. Η Λιθουανία, για παράδειγμα. Το σημαντικό είναι να μπορούν τα κράτη-μέλη ε, να κρατήσουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί ε, ή θα πρέπει, αν χρειαστεί αναθεώρηση, τουλάχιστον να έχουμε μία μεταβατική περίοδο. Γιατί ε, κάποια θερμοκήπια μου είπα στη Λουθανία ότι θέλουν να ε, στραφούν προς τη βιολογική γεωργία, αλλά θέλουν πιο παρατεταμένη μεταβατική περίοδο σε τέτοια περίπτωση. Ε, παρακαλώ, αφήστε τις ευχαριστίες τώρα προς τον κύριο Χόισλινγκ. Αν έχετε να πείτε κάτι ουσιαστικό, καλώς. Αλλιώς θα μην χάνουμε το χρόνο. Σε ευχαριστίες μόνο. Ο κύριος Χόισλινγκ. Λοιπόν, για το ζήτημα των εισαγωγών, εν συντομία, χρειαζόμαστε τις εισαγωγές, όλοι το γνωρίζουμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούνται οι κανόνες ε, και για τις εισαγωγές ε, στο ίδιο επίπεδο όπως και για τους χώρους παραγωγούς. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε όλα αυτά τα διαφορετικά πρότυπα. Αυτό δεν λειτουργεί. Πρέπει να ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλους. Τώρα, το θέμα είναι πώς βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση. Ε, κοιτάξτε τώρα, κύριε Ταραμπέλα, ας μην ξανανοίγουμε μια συζήτηση που έχουμε ήδη κλείσει. Έχουμε ψηφίσει ήδη μια θέση. Ξέρω ότι δεν ήταν όλοι ικανοποιημένοι με αυτή τη θέση, αλλά έχουμε και μια εκστρατεία στον τύπο όπου λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να επιτρέψει τα φυτοφάρμακα στη ε, προϊόντα με βιολογικές ετικέτες. Δεν είναι σωστό αυτό. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα κριτήρια και δεν είναι δίκαιο να υπάρχουν τέτοιου είδου εκστρατείε ε, στον τύπο και να μα παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Ούτε εμεί, ούτε το Συμβούλιο θέλουμε φυτοφάρμακα σε ζωοτροφέ και τρόφιμα. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι αν σε τελική ανάλυση η βιολογική παραγωγή θα πληρώνει το τίμημα για τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι γειτονέ του. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τις προφυλάξεις. Δεν θέλουμε φυτοφάρμακα σε βιολογικά τρόφιμα, αλλά όσον αφορά τα ε, ισοριακές τιμές ή όχι, είναι κάτι που υπάρχει ήδη, το έχουμε ήδη ορίσει και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, οπότε μην ξανανοίγουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Να με συμπαθάτε δεν έδωσα σε όλους το λόγο. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ όμως πολύ σύντομα, τηλεγραφικά. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Χόισλινγκ που είναι ο αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις. Αν έχετε κάτι ειδικό να πείτε, καλώς. Αλλιώς δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια γενικά σχόλια εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά μια σκέψη. Όπως γνωρίζετε και επιθέμησε ήδη ο κύριος Χόισλινγκ, μέχρι στιγμής έχουν λάβει χώρα τέσσερις ε, τριμές διαλόγοι και έπεται πέμπτος. Οι δύο οργανικές διαδικασίες προχωρούν αλλά με αργή ταχύτητα. Η Κομισιόν εκτιμά τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου και της Προεδρίας για την επίτευξη συμβιβασμού σε αυτό το θέμα που είναι πολύ τεχνικής ε, φύσης αλλά και πολιτικά περίπλοκο. Αλλά για να τηρήσουμε τους χρόνους και τις προθεσμίες που προτείνουν η Ολλανδική Προεδρία για να επιτύχουμε δηλαδή η πολιτική συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο, στο τέλος της Ολλανδικής Προεδρίας, πρέπει να επιταχυνθούν οι συζητήσεις. Σε λίγες μέρες, όπως ξέρετε, συμπληρώνονται δύο έτη από την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για αναθεώρηση του κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα. Και αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος ε, να παρεμποδίσει τους βουλικούς παραγωγούς να αναπτύξουν τις πλήρες δυνατότητες τους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ενώ οι ε, επιφάνειες ε, ε, βιολογικής παραγωγής στην Ευρώπη δεν αυξάνονται με την ίδια ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται ευκαιρίες από για τους βιολογικούς παραγωγούς, οπότε πρέπει να επιταχυνθεί η διοργανική διαδικασία ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία μέχρι τα τελή Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας είπα αν έχετε κάτι ειδικό να πείτε. Γιατί σε αυτή τη φάση δεν έχει νόημα να έχουμε σχολιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Τηλεγραφικά. Δεν μπορούμε έτσι να διαχειριστούμε το χρόνο αν παρατείνουμε τη συζήτηση για κάθε θέμα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αποφασίσετε εσεί αν είναι χρήσιμη η παρέμβασή μου ή όχι. Δεν ξέρω αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα μετάφραση, αλλά δεν μπορείτε να μα λέτε ε, εδώ στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου κάτι τέτοιο. Ε, αν έχουμε καθυστερήσει, κύριε Πρόεδρε, αυτό οφείλεται στο ότι δυσκολευτήκατε πάρα πολύ στη διάρκεια τη ψηφοφορία. Οπότε και εσεί πρέπει να δείτε, ε, να γνωρίζετε καλά του καταλόγους ψηφοφοριών. Δεν, δεν μπορούμε να περνάμε σε κάθε ψηφοφορία πάνω από μια ώρα για να ψηφίζουμε ένα κατάλογο ψηφοφορία αρκετά απλό μετά. Αποκλείεται εγώ να μιλάω μετά την Κομισιόν. Η Κομισιόν είναι ένας οργανισμός μη ερετός, ενώ εμείς είμαστε εκπρόσωποι του, των λαών και του γεωργικού κόσμου. Θα κάνετε λοιπόν ό,τι θέλετε, αλλά το πρώτο σας μέλημα πρέπει να είναι να σέβεστε τη δημοκρατία. Αυτό είναι σημαντικό για να μπορούν να εκφράζονται όλοι ελεύθερα. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο. Ε, καλώς λαμβάνω υπόψη αλλά ε, μπας περιπτώσει το σημειώνω παρόλο που δεν ήταν επί της ουσίας το σχόλιο σας. Το λαμβάνω πάντως υπόψη. Περνάμε στο σημείο 10, την έκθεση πρόοδου για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Πρόκειται για γνωμοδότηση του κυρίου Μπόγκοβιτς. Ε, θα σας ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων αν δεν ε, ε, μιλώσετε παραπάνω από ένα πεντάλεπτο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση πρόοδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκπονήθηκε και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά... Και με την έκθεση αυτή ξεκινήσαμε πολύ αργά, διότι έπρεπε πρώτα να δούμε πώς θα γινόταν η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα. Αρχές Φεβρουαρίου υποτίθεται ότι θα γινόταν συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, αλλά αυτό δεν ε, μπόρεσε να γίνει. Ζητώ συγγνώμη. Τώρα έχουν τελειώσει τα προβλήματα και θα θέλαμε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα της ε, Ήτρε. Ήταν πολύ δύσκολο να εκπονήσουμε τόσο γρήγορα μια γνωμοδότηση. Ε, προσλέπω όμως στη μελλοντική συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Είναι σημαντικό το έγγραφο της Επιτροπής, διότι ε, στη το τι θα πρέπει να γίνει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία καθόριζε κάποια μέτρα ε, που θα έπρεπε να ε, εφαρμοστούν μέχρι το 2020. Ε, το 10% των μεταφορών να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να υπάρχουν δεσμευτικές, δεσμευτικοί στόχοι για τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θεσπίστηκαν το 2009. 19 κράτη-μέλη ήδη έχουν ξεπεράσει τους στόχους που είχαν θεσπιστεί τότε. Κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει ακόμα να σημειώσουν πρόοδο για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά ε, ο βασικός στόχος ε, το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανέσιμες πηγές ε, θα μπορέσει να τηρηθεί. Όσον αφορά τις μεταφορές όμως είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Ο στόχος είναι 10% αλλά αυτή τη στιγμή κινούμαστε γύρω στο 6%. Κάτι που βρίσκεται αρκετά κάτω από τον στόχο. Η γνωμοδότησή μας επικεντρώνεται στην γεωργία φυσικά και στην γνωμοδότησή μου δεν είχα πολύ χώρο αλλά αναφέρομαι κυρίως στην στερεά βιομάζα, τα βιοκαύσιμα για τις μεταφορές και την βιοεθανόλη που παράγεται από πρώτες ύλες που είναι γεωργικά προϊόντα ή γεωργικά απόβλητα. Ε, είναι σημαντική πηγή ε, αυτή όμως και μέχρι το 2020 περιμένουμε αυξημένη ζήτηση ε, της βιομάζας σε σχέση με το 2012 27% παραπάνω. Επίσης, Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή των πέλετς θα αυξηθεί από 15 σε 30 ε, ε, εκατομμύρια τόνους. Ε, και η κυρία Κέρστιγκερ ήδη έχει εκπονήσει έκθεση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες από την διαχείριση των δασών. Ε, μπορούμε λοιπόν ε, να, με σωστή διαχείριση να κερδίσουμε πολλά τα δάση χωρίς ε, να τα θέσουμε σε κίνδυνο. Το 75% των πρώτων υλών για τα βιοκάψιμα προέρχεται από εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ζαχαρότευτλα, αραβόσιτο κλπ. Η βιοεθανόλη είναι μια πρόσθετη παραγωγή για την γεωργία. Για τα βιοκαύσιμα όμως ε, χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Στην γνωμοδότησή μου λέω ότι ε, όπως έχει ήδη υποθεί έχει έρθει η ώρα, διότι έχουμε υπερπαραγωγή κάποιων προϊόντων όπως είναι το σιτάρι, τα ζαχαρότεστλα και ο αραβόσιτος. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα ε, προϊόντα αυτά για την παραγωγή βιοεθανόλης. Με την κατάργηση των ποσοστώσεων της ζάχαρης υπάρχει υπερπαραγωγή ε, ζαχαρότευτλων. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό. 20 Απριλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και 25-26 θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές και θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να συμφωνήσουμε όσον αφορά τις τροπολογίες. Βιαζόμαστε λόγω του χρονοδιαγράμματος της Ήτρε όπου θα συζητηθούν οι τροπολογίες στις 20 Απριλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που εμείνατε και στο χρόνο το σύντομο που είχατε. Κύριο Καπούτο, σύντομα παρακαλώ κι εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο εισηγητής ο κ. Μποκοβίτς ε, παρουσίασε ήδη τις ε, οργανωτικές και τεχνικές δυσκολίες που μας εμπόδισε να κάνουμε μια συζήτηση πιο πλήρη. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Υπάρχει όντω ανάγκη οι ανανεώσιμε πηγέ ε, βιολογικών ενεργειών να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα τη ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη μπορούν επίσης ε, να αποτελέσουν και όθηση για, αυτή την, ε, για την οικονομία και την κοινοτομία στην Ευρώπη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στον τομέα της γεωργίας μπορούν να προγραμματιστούν και αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μια δυνατότητα σταθεροποίησης του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθούν η έκθεση πιστεύω θα έπρεπε να περιλαμβάνει και μια αναφορά στα έξυπνα δίκτυα, στα smart grids, τα οποία θα επιτρέψουν πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανενώσιμων πηγών ενέργειας γεωργικής προέλευσης. Απομένουν και υπάρχουν ακόμα διάφορα κανονιστικά εμπόδια και εμπόδια στις αγορές των κρατών μελών, σημαντικά εμπόδια για την ανάπτυξη των smart grids, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ε, μέχρι τα κράτη-μέλη να καταφέρουν να καταργήσουν, να άρουν αυτά τα εμπόδια. Μια άλλη πτυχή, ε, ενώ κατά τα συμφωνώ με τον εισηγητή, μια άλλη πτυχή που πιστεύω πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση είναι η αναφορά στις ε, αγροενεργειακές περιοχές όπως ονομάζονται που θα επιτρέψουν ε, την παραγωγή βάσει ε, αποβλήτων της γεωργίας. Όπως ξέρουμε αυτές οι ενεργειακές περιοχές ε, θα αποτελούν εδαφικές ενότητες που θα συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες ικανότητες για τις ενδιάμεσες φάσεις μεταξύ της παραγωγής της ενέργειας και της διανομής της πρόβλεψη λοιπόν κινήτρων εκεί για τα κράτη-μέλη ώστε να αναπτύξουν αυτές τις περιοχές ε, κατά την άποψή μου θα ήταν επιθυμητή. Ο κύριος Αντρέα παρακαλώ να είστε λακωνικός κι εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σημαντικό είναι στην γνωμοδότηση αυτή να κάνουμε κάποια σχετικοποίηση. Ο συντάκτης γνωμοδότησης ε, περιορίζει τη βιομάζα στις καλλιέργειες και στο ξύλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε, αλλά να μιλήσουμε και για τα απορρίμματα της βιομάζας και τα υποπροϊόντα των καλλιεργειών. Γιατί η συζήτηση είναι ίδια. Αν δεν ε, προσέξουμε, ε, ίσως ε, υπάρξει μια σύγκρουση μεταξύ των καυσίμων και των ε, ε, τροφίμων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προβληματιστούμε γι' αυτό. Επίσης, η απόδοση του κλάδου των βιοκαυσίμων. γιατί ξέρουμε ότι τα, καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα ε, πολλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ διαρθρωτικής κατάστασης και συγκυριακής. Επίσης, έχουμε και τις γεωργικές πρώτες σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάτι που ερχόμαστε σε αντίφαση γιατί για να ε, διαφυλάξουν το γεωργικό τους εισόδημα χρειάζεται να αυξήσουν την παραγωγή τους. Αλλά έχουν ε, μια στασιμότητα και στην απόδοση δυστυχώς. Ταυτόχρονα έχουμε και το πρόβλημα της σημερινής κρίσης ε, και την ανάγκη να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα της ιωρικής παραγωγής. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ με τον εισηγητή να προωθήσουμε τους ε, τοπικούς συνεταιρισμούς ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επίσης η ανάπτυξη μεμονωμένων ή συλλογικών σχεδίων στην Ήπεθρο δίνουν δυνατότητα διαφοροποίησης του γεωρικού εισόδηματο μία διαφοροποίηση λοιπόν είναι σημαντική, αλλά με προσοχή και σύνεση. Επίσης, να δούμε τι μέσα έχουμε στην ε, πολιτική της ανάπτυξης για να ενισχύσουμε προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αν θέλετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε κάτι καινούργιο, να μην επαναλαμβάνετε σχόλια που έχουν ήδη γίνει. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, η γνωμοδότηση αυτή, πολύ σημαντική και για τη Γεωργία, γιατί θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε την υπεθρό μας και ευρύτερες ε, περιοχές ε, γιατί υπάρχουν περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ε, ε, μεγάλο, μεγάλη παραγωγή βιομάζας ε, που ξεπερνά τις εθνικές ανάγκες. Είναι σε μερικές φορές. Και επίσης η βιωσιμότητα είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο. Ας μην ξεχνούμε σήμερα, ότι σήμερα ε, αγοράζουμε το 50% των ενεργειακών προϊόντων που χρειαζόμαστε 400 δισεκατομμύρια το χρόνο δαπανούμε σε εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων. Και θα μπορούσαμε αυτά τα κονδύλια να τα αξιοποιήσουμε, αυτά τα χρήματα να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα από το να εισάγουμε συνεχώ ενεργειακά προϊόντα. Οπότε η βιοενέργεια θα μπορούσε όχι μόνο να αυξήσει το γεωρικό εισόδημα των παραγωγών, αλλά να γεμίσει και τα δημόσια ταμεία. Και η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοαέριο, όχι μόνο για τη θέρμανση ή για βιοκαύσιμα. Έτσι θα μειώσουμε και την ρήπανση. Και μην ξεχνάτε και τα απορρίμματα από, το, από την υλοτομία και πόσο ξύλο πάει χαμένο γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά. Και αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων. Ο κύριος Ελιμόβιτς. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόγκοβιτς για την ε, εξαιρετική του γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και να εκφράσω τη συμφωνία μου με τα περισσότερα τμήματά της. Εδώ θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη εξυγχρονισμού της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη για να καταφέρει να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες ε, της γεωργίας των περιβάλλων και να συμβάλλει σε αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η γνωμοδότηση αναγνωρίζει ότι ο τομέας των μεταφορών δεν έχει καταφέρει ε, να τηρήσει το στόχο το 10% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε και να βρούμε νέες λύσεις. Και όταν μιλούμε για τις μεταφορές, να μην ξεχνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για ηλεκτρικά οχήματα, όχι μόνο βιοκαύσιμα, για να έχουμε όλο και πιο φιλοπεριβαλλοντικά καύσιμα. Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχής αφορά τις υποδομές. Χρειαζόμαστε υποδομές για τη μεταφορά όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράγουμε στην Ευρώπη γιατί σε μερικέ χώρε έχουμε μεγάλη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, αλλά αν δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε σε άλλε χώρε που δεν παράγουν τόσο πολύ, τότε προστεί αυτή, αυτό το πλεόνασμα παραγωγής σε ορισμένες χώρες. Επίσης, ένα αντιφατικό, επίμαχο μάλλον ζήτημα, το Nord Stream 2. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχα περισσότερο χρόνο. Πιστεύω ότι τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ενεργειακή παραγωγή. Οπότε δεν συμφωνώ με την παράγραφο 6 της ε, γνωμοδότησης, αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που διάβασα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία υπάρχει μια προσπάθεια να φυτεύονται περισσότερα δέντρα ως ενεργειακή πηγή, αλλά ένας τομέας που θα πρέπει να εξετάσουμε δεν ξέρω τι γίνεται στο υπόλοιπο της Ευρώπης, ε, ε, χρησιμοποιούνται οι βάλτοι. Ε, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν πολύ καλά, βλάπτουν τους βάλτους, εκπέμπεται μεθάνιο στην ατμόσφαιρα και καταστρέφονται περιοχές που βοηθούν στο μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Παρότι λοιπόν δεν έχει πολύ νόημα αυτή η προσπάθεια, φαίνεται να προχωράει. Θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και επίσης, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα για το αυτοκίνητό μου, ε, ε, μου είναι δύσκολο να οδηγώ το αυτοκίνητό μου με βιοκαύσιμα που έχουν παραχθεί από τρόφιμα τη στιγμή που ακούω στο ραδιόφωνο ότι ο κόσμο στην Αφρική πεθαίνει από την πείνα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλό που συζητάμε τι διάφορε ανάμεσα στι διάφορε χώρε. Ε, υπάρχουν ε, σημαντικές διαφορές. Ε, κάποιες χώρες έχουν προοδεύσει περισσότερο από άλλες. Νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε τις μακροπρόθεσμες λύσεις. Την έρευνα για παράδειγμα, διότι βλέπουμε ότι χρησιμοποιώντας εκτάσεις για το στην ε, Δανία και στην ε, Γερμανία ε, πληρώνει κανείς ενίκιο για την έκταση αυτή, εξωθούνται κάποιοι γεωργοί, υπάρχουν λοιπόν συνέπειες από τις επιλογές αυτές. Από την άλλη η έρευνα μπορεί να Ε, μας βοηθήσει, για παράδειγμα, την αιωλική ενέργεια που παράγεται και που δεν χρησιμοποιείται να την ε, μετατρέψουμε σε υδρογόνο για ε, χρήση σε αυτοκίνητα και στον τομέα των μεταφορών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες, αλλά ιδιαίτερα την έρευνα και τις μακροπρόθεσμες λύσεις, ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ευχαριστώ. Pani poseł Ευχαριστώ κύριε Νταμάτο. Η Νταμάτο, συγγνώμη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης επικεντρώνεται κυρίως στα βιοκαύσιμα. Ο εισηγητής ε, μας το είπε για λόγους συντομίας. Αλλά ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ανανοησιμές πηγές ενέργειας ε, αναφερόμαστε και στην ηλιακή, στη γεωθερμία και στην ε, σε άλλες μορφές παραγωγής ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την καύση των ε, αποβλήτων και τους στόχους που πρέπει να επιτύχουμε μέχρι το 2020, δηλαδή το 20% σε εναλλακτικέ ε, μορφές ενέργειας. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το μοντέλο εξάρτησης από τα ρεκτά καύσιμα με ένα άλλο το οποίο θα ασχολείται με όλες τις μεγάλες πολυεθνικές ε, που ασχολούνται με τις ε, μορφές η ενέργειας, ε, ηλιακής ενέργειας, επιβάλλοντας τιμές δικές τους. Πρέπει να διευκολύνουμε τη χρήση της γης με την επάρκεια ενεργειακή, επάρκεια και βάζοντας στο δίκτυο το πλεόνασμα της παραγωγής ε, η γη δεν είναι κάτι ε, που δεν εξαντλείται. Ε, χρειάζονται πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί μια γη μετά από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Το ίδιο και όταν χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά πάνελ. Κάθε απόφαση επηρεάζει την παραγωγή τροφίμων και τη γη πολλές ε, βλάβες ε, ε, δημιουργούνται από διάφορες μορφές παραγωγής ενέργειας. Εμείς θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να εισάγουμε αυτές τις βελτιώσεις. Ευχαριστώ κύριο Άγνιου. Ευχαριστώ. Μιλούμε για τη βιομάζα, κυρίως ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και διαρωτάμε αν η γραμμοδότηση επισημαίνει πόσο έφερα στην η κατάσταση αυτή. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε μεγάλες αποστάσεις ε, ε, χάνουμε πολλά κονδύλια. Το έχω βιώσει και προσωπικά. Δύο βασικά στοιχεία είναι που ισχύει για τη βιομάζα. Πρέπει να είναι τοπική χρήση και η παραγωγή δεν θα πρέπει να είναι δαπανηρή. Μόνο έτσι είναι βιώσιμη η παραγωγή βιομάζας. Αλλιώς χάνουμε χρήματα. Ένα άλλο σημαντικό για τη βιομάζα είναι όταν πηγαίνουν σιτηρά σε ένα εργοστάσιο εθανόλης, αφαιρείται η εθανόλη για το καύσιμο και αυτό που απομένει είναι χρήσιμη ζωοτροφή, είναι πρωτενη. Και έτσι γλιτώνουμε και από τις αγωγές της σόγιας. Αυτό δεν αναφέρεται γιατί είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπο τρόπος για βιομάζα μεγάλη κλίμακος μάλιστα. Ευχαριστώ. Κυρία Πετήρ επιμένετε ή δεν χρειάζεται. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπόγκοβιτς για την πολύ αξιόλογη γνωμοδότηση, τον συγχαίρω για τις προτάσεις του. Πολύ σωστά επισήμανε την, το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για τη γεωργία και τις αρμοδιότητες επιτροπής μας. Ε, αναφέρθηκαν κάποια θέματα που άπτονται και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και σίγουρα αυτές τις προτάσεις θα τις μεταφέρουμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι πάντως σημαντικό, ε, είναι σημαντική η γεωργική έκταση και μάλιστα γεωργικές εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται. Γιατί υπάρχουν τέτοιες καλλιέργητες γεωργικές εκτάσεις σε πολλές χώρες και κυρίως στις νέες χώρες. Θα πρέπει αυτές οι γεωργικές γεές να αξιοποιηθούν προς το συμφέρον τοπικού πληθυσμού και οι πρώτες ύλες που παράγονται εκεί να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή βιοκαυσίμων. Και εκεί δυστυχώς υστερούμε σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ε, θα πρέπει να, στηρίξουμε, να και την ε, ε, ανάπτυξη της δασοκομείας που περιορίζει και την περιβαλλοντική ρήπαση αλλά και αυξάνει την παραγωγή βιομάζας. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές και τους στόχους που έχουμε θέσει για αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε την αργή πρόοδο σε σχέση με την γραφειοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διατυπώσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τζούλιο Βάλπη, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, να κάνει μια σύντομη όμως τον θέρμα παρακαλώ παρέμβαση. Yes, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επικροτούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που ακούσαμε. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή μας έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο η Ευρώπη ε, να κατέχει ηγετική θέση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και ε, αυτό, θα θεσπι... αυτό θα επιτευχθεί με την επίτευξη του στόχου του 20% του 2020 ε, και του 27% του 2030. Να θεωρούμε λοιπόν την ε, οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να θεσπίσουμε το πλαίσιο για το 2030. Επίσης, όπως ακούσαμε, θα πρέπει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, να ενσωματωθούν στο ενεργειακό μας σύστημα. Η βιοενέργεια λοιπόν μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί ε, στο θέμα αυτό, διότι είναι πολύ ευέλικτη μορφή ενέργειας. Μπορεί να παράσχει θέρμανση, ε, ρεύμα και να χρησιμοποιηθεί στις μεταφορές. Ε, θα είναι χρήσιμο λοιπόν να υπάρξουν ε, ε, συνεταιρισμοί και επίσης να προωθήσουμε τα μέτρα για απαλλαγή των μεταφορών από ανθρακούχες εκπομπές. Τέλος, ως μέρος της αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για μετά το 2020, εξετάζουμε και την ενδεχόμενη αναθεώρηση της πολιτικής βιωσιμότητας για την βιοενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξετάσουμε λοιπόν και τα βιοκαύσιμα αλλά και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την βιώσιμη διαχείριση των δασών και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες όπως είναι ο ανταγωνισμός του τομέα τροφίμων με τον τομέα των καυσίμων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει ο κύριος Μπόκοβιτς να δευτερολογήσει. Παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ και για την κατανόησή σας ε, που δεν μπορέσαμε ακόμα να οργανώσουμε ε, συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές. 22 Μαρτίου λοιπόν είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Είναι σαφές τώρα το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ε, προτάσεις που μας υποβάλλατε μέχρι τώρα. Βλέπουμε σημαντική αστάθεια των τιμών, για παράδειγμα στο πετρέλαιο και στόχος μας θα πρέπει να είναι ε, να έχουμε πιο σταθερό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα. Η γεωργία λοιπόν ε, μπορεί να οδηγήσει σε εξειδίκευση και στο σημείο 6 έχουμε κάπως ε, αγωνιστικό ύφο εκεί που μιλάμε για μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών. Αλλά και στο γάλα συνέβη το ίδιο. Όταν καταργήθηκαν οι κανόνες ε, ε, και για τη ζάχαρη το 2016-2017 θα δούμε το ίδιο. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε το θέμα της, ε, ε, του πλεονάσματος ε, στην παραγωγή. Το θέμα αυτό λοιπόν συνδέεται και με στόχους φιλικούς προς το περιβάλλον και υπάρχουν ακαλλιέργητες εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, όπως ε, και η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια. Εάν έχουμε λοιπόν ε, παρόμοια ρύθμιση και στον τομέα της γεωργίας ε, θα Έχουμε και εκεί μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών. Προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων. Ω συντάκτη τη νομοδότηση έπρεπε να περιοριστώ στην ε, γεωργία και φυσικά ε, είχα και περιορισμό όσον αφορά το μήκο ε, τη νομοδότηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Πώς να εξηγήσω στον συνάδελφο ότι είχε λίγο χρόνο. Γιατί πάντα μας λείπει χρόνος για τα πολύ σημαντικά θέματα και όλες οι συζητήσεις παρατείνονται, αλλά ειδικά για τα πολύ σημαντικά θέματα δεν μπορώ να περικόπτω το χρόνο. Λοιπόν, περάμε στο θέμα της αστάθειας των τιμών. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας κάνει την ενημέρωση. Merci, Monsieur Κύριε Ντελαέ. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Αν και όπως είπα το θέμα είναι πολύ σημαντικό και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άλλες συζητήσεις για το ίδιο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της βαθύτατης κρίσης που βιώνει αυτή τη στιγμή. Η αστάθεια των τιμών, οι απότομε διακοιμάσει έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Και παρόλο που οι διακοιμάσει είναι γενεί οποιοδήποτε μηχανισμού αγορά, τόσο σημαντικέ διακοιμάσει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι ένα έκτακτο φαινόμενο. Και το φαινόμενο αυτό φυσικά ε, έχει κάποιε συνέπειε και για του γεωργού. Αυτή η τεράστια αστάθεια δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα για του γεωργού και δεν μπορούν να κάνουν προβλέψιμες ε, πολιτικές, κάτι που εθαρρύνει και τις κερδοσκοπικές ενέργειες. Τώρα, έχουμε δυστυχώς ένα παγκόσμιο φαινόμενο και επηρεάζει και το σύνολο των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με την κοινή γεωρική πολιτική να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο τη μεγάλη αστάθεια των τιμών. Εμείς ως ε, Ευρωπαίοι νομοθέτες έχουμε ευθύνη να προτείνουμε λύσεις για να βελτιώσουμε το γεωργικό εισόδημα. Στην δημόσια κρόση με πυρογνώμονες το Φεβρουάριο είδαμε να σκιαγραφούνται κάποιες προτάσεις θα σας ε, αναφερθώ στα βασικά. Το σύστημα ασφαλίσεων, οργάνωση σε δύο πυλώνες της κοινή πολιτικής, διαφάνεια των αγορών, άμεσες ενισχύσεις, μέτρα διαχείρισης της κρίσης μέσω προγραμμάτων ε, πρόθεσης και διαφήμιση, αντικυκλικά συστήματα, εμπορικές διαπραγματεύσεις, δίκαιο ανταγωνισμού και τέλος η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του G20. Βέβαια δεν είναι τα μοναδικά θέματα που πραγματευτήκαμε σε αυτή τη δημόσια κρόαση του Φεβρουαρίου με τους εμπειρογνώμονες. Πάντως ε, ανέκυψε τότε ε, ο έντονα τεχνικός αλλά και ο ιδιαίτερα πολιτικός χαρακτήρας του θέματος της αστάθειας των τιμών. Και φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, ως επαγγελματίας γεωργός δεν ενδιαφέρομαι για την βιβλιογραφία αλλά για συγκεκριμένα και χρήσιμα αποτελεσματικά μέτρα για τους γεωργούς. Χρειαζόμαστε σαφή απλά και ακριβή μέτρα, γιατί πολλά περιμένουν από από εμά η Γεωργή και η παρούσα συγκυρία μας υποχρεώνει σε έναν ρεαλισμό. Προσπαθώ με την έκθεση αυτή να προσφέρω στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες ε, σκέψεις ε, και προτάσεις λύσεων, ώστε η απάντηση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2020 είναι ακόμη πιο αποτελεσματική. Η έκθεση περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Το Η πρώτο είναι μια αντικειμενική διάγνωση του φαινομένου της αστάθειας των τιμών και των συνεπειών που έχει αυτή η αστάθεια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο δεύτερος άξονας ε, προσδιορίζει τους στόχους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και προτείνει και μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική και τρίτον προτάσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανέβρεση λύσεων. Θα μπορούσα ήδη να σας αναφέρω τους ε, στόχους που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικοί. Τρεις είναι οι βασικοί. Η επιστημιστική κυριαρχία της Ευρώπης, η βιωσιμότητα των ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση των βιωτικών συνθήκων των γεωργών. Και ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία για καρποφόρα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Και θα ήθελα να έχει θετική απήχηση και στο γεωργικό κόσμο αυτή η έκθεση, γιατί αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί ε, ο γεωργικός πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τους, εκ των τους και οδησηγητές. Εγώ πρόκειται να συντάξω την έκθεση έχοντας δώσει προηγουμένως την ευκαιρία σε όλους τους συναδέλφους να καταθέσουν τις απόψεις και να ε, στηρίξουν τα επιχειρήματά τους. Είμαι ανοιχτή και περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια και τις απόψεις. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Περάμε στη συζήτηση και θα έλεγα Όποιος έχει προτάσεις να τις ε, υποβάλει και προσωπικά στην εισηγητρία και διμερός ε, και θα έχουμε και την ε, ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της συζήτηση των τροπολογιών. Εγώ έτσι, μέσω τροπολογιών υποβάλλω τις προτάσεις μου στις διάφορες εκθέσεις. κυρία Μίλλερ. κυρία Μίλλερ, παρακαλώ. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της γενικής κατεύθυνσης που θα μας πάει το ταξίδι αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αστάθεια των τιμών. Για μένα δύο πράγματα είναι σημαντικά. Καταρχάς, όσον αφορά τους νέους γεωργούς, να τους προωθήσουμε, να τους δείξουμε ότι έχουν μέλλον. Για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον δεύτερο πυλώνα να συνεχίσουμε να έχουμε ευρύ περιθώριο για τις περιφέρειες. και χαίρομαι ιδιαίτερα που θύμεται κυρίως το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας. Ωστόσο βρίσκω δύσκολο να να συνδυάσουμε τις διάφορες πτυχές, διότι ο τομέας των τροφίμων είναι πάρα πολύ σημαντικός στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε και τις εμπειρίες που έχουμε από το greening, ε, την ε, περιβαλλοντική κατεύθυνση που θα δίνεται. Πιστεύω ότι έτσι τελικά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τη λακωνικότητά σας ιδιαίτερα. Ο κύριος Άγνιου. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετριάσουμε τις συνέπειες της αστάθειας των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Ε, μπορώ να προτείνω και δύο μέσα εδώ πέρα. Έχουμε τις, ε, τις προθεσμιακές ε, αγορές. Ε, συχνά βλέπουμε κόσμο που κερδοσκοπεί στον τομέα αυτών σημαντικό είναι να ε, καλλιεργεί ο γεωργός ε, γνωρίζοντας ε, την τιμή του προϊόντος του ήδη κατά την καλλιέργεια. Με ενοχλεί όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δυσκολέψει όσο γίνεται τις προθεσμιακές αγορές. Και το δεύτερο εργαλείο είναι κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο στον Ηνωμένο Βασίλειο. Οι λιανοπολιτές συνεννοούνται με τους παραγωγούς ε, ώστε ε, αν αυξάνεται η τιμή των ζωοτροφών αυξάνονται αυτομάτως ε, και οι τιμές. Το γνωρίζω αυτό διότι ασχολούμαι ακριβώς με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βατσό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά η αστάθεια των τιμών είναι δραματική για τον γεωργικό κόσμο δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους παραγωγούς και πλήττει τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των εκμεταλλεύσεων. Έχει ξεκινήσει από τις αρχές ε, του 2000 ε, λόγω μερικές φορές ε, σημαντικών και απρόβλεπτων αυξομοιώσεων των τιμών. Ταυτόχρονα η γεωργική πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο ε, για τη γεωργία έχει τεράστιες διαφορές από περιοχή σε περιοχή ε, κατά 70% έχει αυξηθεί η γεωργική παραγωγή ε, στην Αμερική, στην Κίνα, στη Βραζιλία ενώ εδώ έχει μειωθεί. Τα πράγματα λοιπόν είναι σαφή. Ε, όταν ε, αναφέρομαι σε ποσοστώσεις, σε αποθήκευση, σε κανονισμούς ε, όλα αυτά δημιουργήθηκαν υπό την πίεση της ενιαίας οργάνωσης αγοράς. Έτσι λοιπόν οι τιμές ε, ευθυγραμμίστηκαν με τις παγκόσμιες. Οι προθεσμιακές αγορές επίσης ε, ασκούν πιέσεις στη γεωργική παραγωγή. Η γεωργική πολιτική λοιπόν πρέπει να διασφαλίζει επαρκή αμοιβή, ε, διασφάλιση των εισοδημάτων των γεωργών, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να διασφαλίζει τη μακροβιότητα των παραγωγών μας, των καλλιεργιών μας με την αναθεώρηση της ε, κεντρικής, ε, ε, κοινής γεωργικής πολιτικής δεν διαφαίνεται αυτό ο στόχος. Πώς θα γίνει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική ώστε να επανακτήσουν την κυριαρχία τους ή γεωργοί. Ευχαριστώ. Ο Φεράν. Ευχαριστώ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε που στείλατε επιστολή στον Επίτροπο Χόγκαν. Τη διάβασα με μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να στηρίξουμε πολλές παραγράφεις της επιστολής ε, και κυρίως μέσω της Επιτροπής μας. Ο κύριος Λοζό με κάλυψε. Σήμερα δεν έχουμε κανένα πραγματικό μηχανισμό για τη μείωση της αστάθειας των τιμών. Και τα διάφορα πακέτα ζάχαρης, γάλακτος και το καθεξής δεν είναι παρά πλάνες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μόνο ρυθμίση παραγωγής αυτή τη στιγμή με έναν ορθολογικό προστατευτισμό θα μας επέτρεπε να επανέλθουμε σε ένα φυσιολογικό επίπεδο τιμών. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ε, δεν έστειλε επιστροπή στον ε, Επίτροπο Χόβεν, αλλά στον πρόεδρο Γιούνκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια η αστάθεια των τιμών ε, για τα γεωργικά προϊόντα αποτελεί σταθερά, σταθερό κίνδυνο για τους γεωργούς ενώ η Ευρώπη αποδομεί μεγάλο κομμάτι των παραδοσιακών καλλιεργιών και πραγωγών εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά την εισηγήτρια. Συμφωνώ με την προσέγγιση που θέλει να υιοθετήσει σε αυτή την έκθεση. Το θεωρώ θεμελιώδη σημασία, ειδικότερα δεδομένων ε, των συνθηκών ε, του περιβάλλοντος εντό του οποίου συζητάμε. Αλλά θέλω να ανοίξουμε λίγο και τη συζήτηση για, όσον αφορά τι καινοτόμε μορφέ ε, γεωργία. Η γεωργία έχει αλλάξει πλέον. Έχει αλλάξει και το οικονομικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται. Δεν πρέπει λοιπόν να παραβλέπουμε τη δυνατότητα να αναφέρουμε καινοτόμες μεθόδους που ενδεχομένως θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της αστάθειας των δημών Από αυτή την άποψη ε, και στη συζήτηση που είχαμε με τον Επίτροπο Χόγκαν ε, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι πρέπει να μελετήσουμε πιθανές παρεμβάσεις ε, που ενδεχομένως θα δανειστούμε και από τα πράγματα που έγιναν γενικότερα για τη διάσωση του ευρώ, την ποσοτική χαλάρωση, όλα αυτά. Κατά την απόψή μου υπάρχουν τέτοια περιθώρια αν σκεφτεί κανείς και τη δυνατότητα να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με νέους τρόπους αντιμετώπισης. Από αυτή την άποψη λοιπόν ελπίζω μαζί με την εισηγήτρια να καταφέρουμε να εντοπίσουμε μια οδό που θα φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι σημαντικό είναι για να συγυρίσουμε τους κανόνες για τους διάφορους ε, τρόπους επιδότησης. Ε, βλέπουμε ότι η Γαλλία θέλει να αγοράσει τα πλεονάσματα, άλλοι δεν θέλουν. Σημαντικό είναι να έχουμε τις ίδιες συνθήκες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να έχουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Έχουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. αλλά έχουμε μια αγορά που ρυθμίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση και οι ε, τιμές στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει να μας καθοδηγούν και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ε, παράγουμε προϊόντα και ο κόσμος να είναι διατεθειμένος να πληρώσει την τιμή ε, που στοιχίζει το προϊόν. το να εξαγοράζουμε τεράστιες ποσότητες ε, σίτου επειδή ε, έχει, πέσει, ε, έχει ευξηθεί η παγκόσμια παραγωγή κατά 2,3% σημαίνει ότι παράλληλα υπάρχει κάποιος κάπου αλλού που κερδοσκοπεί και οδηγεί σε αύξηση των τιμών κατά 70%. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι ανταγωνιζόμαστε στην διεθνή αγορά και θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης πώς η συμφωνία TTIP θα επηρεάσει τις αγορές μας στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Το θέμα της αστάθειας των τιμών δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ομοιόμορφα, γιατί τα αίτια αύξηση των τιμών χρήζουν τελείως διαφορετικής αντιμετώπισης από τα αίτια απότομη μείωση των τιμών. Γιατί η απότομη μείωση σχετίζεται με την υπερβολική παραγωγή, ενώ η απότομη αύξηση μπορεί να οφείλεται σε ε, ε, ελληματική παραγωγή ή σε δυσλειτουργίες που οδηγούν σε εκτροπές. Οπότε, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο, κάποια βαρύτητα στις διάφορες χώρες και να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών, πρέπει να ε, αναλάβουμε πανευρωπαϊκή δράση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια στο G20 και στη ΦΑΟ. Ήδη η, ομάδα των G20 έχει ξεκινήσει μια προεργασία, αλλά εδώ και καιρό έχει εξαφανιστεί από τις προτεραιότητες, ενώ η ΦΑΟ ε, θα πρέπει να συνεχίσει τις ε, μελέτες της ε, και καλό θα ήταν να έχουμε και μία κρόση με εκπροσώπους στη ΦΑΟ για να δούμε σε τι συμπεράσματα έχει καταλήξει. Αν ε, καταφέρουμε να ελέγξουμε τις απότομες διακοιμάνσεις σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να βρούμε μετά κάποιες εσωτερικές προσαρμογές. Έχουμε διάφορους μηχανισμούς παντού και στην Ευρώπη μέσω των διαφόρων μορφών ασφαλίσεων για παράδειγμα ώστε να αποφύγουμε μόνο με εσωτερικέ αποφάσεις να λύσουμε ένα πρόβλημα που είναι θέμα μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να τονίσω αυτά που υπόθηκαν, ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Νταντάν. Στην Γερμανία όταν ε, συναντιέμαι με γεωργούς, Ε, μου μιλάνε συχνά για ε, τις εθνικές αρμοδιότητες. Ε, θα πρέπει να υπάρξει φορολογική ρύθμιση και για τη, τους γεωργούς. Δηλαδή, ε, όταν έχουν καλή σοδιά να πληρώνουν υψηλούς φόρους, αλλά αντίστροφα όταν η χρονιά περάσει λιγότερο καλά να πληρώνουν μειωμένους φόρους. Όσον αφορά τη ρύθμιση των ποσοτήτων, θα ήθελα να πω ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργήσει μόνο αν ε, έχουμε και προστασία, διότι αν ε, δεν το έχουμε αυτό, δεν θα λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ευφιέστερα συστήματα, διότι με το παρόν ως έχει δεν θα μπορέσουμε να πληροφορήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Χανιώτη, τον εκπρόσωπο, το Διευθυντή και τον εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μας παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ κύριε Χανιώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να εξηγήσω ευθύ εξ αρχή ένα πράγμα. Θέλουμε η συνεργασία μας με τον εισηγητή να είναι όσο το δυνατόν εκτενέστερη. Έχουμε στείλει ήδη κάποιε πληροφορίε ε, που προκύπτουν από παλαιότερε αναλύσει που έχουμε κάνει στον τομέα. Επικαιροποιούμε τώρα τι αναλύσει όλων των διαθέσιμων μέσων βάσει των νέων επιπεδοτημών και φυσικά είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε οποιασδήποτε διευκρινήσεις ε, να δώσουμε οποιασδήποτε διευκρινήσεις ε, θα ήθελε ο εισηγητή σας η επιτροπή σας επίσης θα ήθελα να εξηγήσω ένα-δυο άλλα πράγματα τα οποία ίσως να μην έγιναν σαφή με την προηγούμενη μου παρέμβαση στην ακρόαση που είχε γίνει δεν θα μιλήσω για το στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις προτάσεις της Κομισιόν ε, όσον αφορά τι προτάσει τη Κομισιόν. Αυτό είναι δική σα αρμοδιότητα. Θα επικεντρωθώ στην αντικειμενικότητα των γεγονότων και θα προσπαθήσω να τονίσω για άλλη μια φορά ένα στοιχείο το οποίο μας φαίνεται ότι δημιουργεί σύγχυση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε τη Γεωργία υπό ε, μια ρόδινη εικόνα. Είναι σαφές ότι όταν πέφτουν ή ανεβαίνουν οι τιμές η Γεωργία αντιμετωπίζει πάντα τα ίδια προβλήματα οι τιμές ε, των γεωργικών προϊόντων αυξάνονται μόνο κατά το 1 δέκατο σε σχέση με το τι συμβαίνει στα λοιπάσματα και στην ενέργεια και όταν πέφτουν το ίδιο συμβαίνει πάλι. Μιλάμε λοιπόν για ένα φαινόμενο το οποίο από τεχνική άποψη ονομάζεται υποβάθμιση των όρων συναλλαγών πρακτικά σημαίνει ότι οι γεωργοί ε, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κόστους. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι η αβεβαιότητα των τιμών είναι το σημαντικότερο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Όταν έχουμε μια μέση τιμή 100 ευρώ όπως συνέβαινε με τα δημητριακά για δεκαετίες και ξαφνικά ανέβουν οι τιμές κατά 20 ευρώ ή πέσουν κατά 20 ευρώ ε, μπορεί κανείς να δει την τάση και την αστάθεια, μπορεί να την μετρήσει. Αλλά όταν σε ε, μια οκταετία ε, δύο φορές ανεβαίνουν και δύο φορές καταραίουν οι τιμές, πάβει να υπάρχει τάση και δεν μπορεί κανείς να ε, μετρήσει την αστάθεια. Για να τα πω λοιπόν συντομία, υπάρχουν τρεις παράλληλες εξελίξεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η αστάθεια, η αβεβαιότητα των τιμών και η παράλληλη εξέλιξη αυτή και αυτά μας δημιουργεί πρόβλημα αν εστιαστούμε πλέον και στις τρεις λύσεις. Αλλά αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και θα σας παρέχουμε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στις δικές σας συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που υπόσχεστε να μας υποστηρίξετε. Θα παρακαλούσα την εισηγήτρια να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, διότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες για τη συμμετοχή τους. Ε, τα σημείωσα όλα και θέλω να ακούσω τα σχόλιά τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ε, διότι το χρονοδιάγραμμα είναι λίγο πιεσμένο. Εγώ έχω προβλέψει να στείλω προς μετάφραση περίπου 20 Απριλίου την έκθεση, δηλαδή πρέπει να είμαστε αρκετά γρήγοροι. Θα ήθελα να καθισκάσω την Κομισιόν. Πράγματι θα γίνει διάλογος μεταξύ εισηγητρίας και σκιωδών και ε, θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι όλοι θέλουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων Γεωργών οπότε είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε λύσεις για να προστατεύσουμε τον Ευρωπαίο Γεωργό για το μέλλον και να προετοιμάσουμε την επόμενη κοινή πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντελαέ. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και τις ε, εθνικές εμπειρίες. Είχαμε τον Ισπανό Υπουργό Γεωργίας που μας μίλησε για αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε κάποια κατακαιρματισμένη προσέγγιση και εθνικές εμπειρίες, το ανέφερε και ο κύριο Άγνιου. Αυτό το γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν αξιοποιήσετε λοιπόν και τις εθνικές εμπειρίες θα εμπλουτίσετε αυτή την πολύ σημαντική και δύσκολη έκθεση. Σας ευχόμαστε καλή τύχη, καλή επιτυχία. Σίγουρα θα έχουμε και δεύτερη ανταλλαγή απόψεων αφού ολοκληρωθούν και οι μεταφράσεις ε, του σχέδιου έκθεσης και θα επανέλθουμε. Ένα δίλεπτο διακοπή τεχνική και μετά θα περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων το θυρών. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα μόνο οι συντονιστές παρακαλώ να παραμείνουν στην αίθουσα.